Pan Κυρίες και κύριοι, ε, ξεκινάμε λοιπόν και πριν προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης, θα ήθελα να μου να κάνω μια σύντομη δήλωση η γραπτή δήλωση η 45 κάθετος 2011